Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τα προφορικά ερωτήματα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα την ερώτηση με έτοιμα προφορική απάντηση για το πρόγραμμα Ευθύ Ενέργεια στην Ευρώπη. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την πρώτη εισηγήτρια τη ερώτηση, την κυρία Καρβάλιο, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κατά πρώτον ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να θέσω αυτή την ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνέχιση του προγράμματος ευφυής ενέργειας στην Ευρώπη. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν πολύ, σημαντική, πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει στρατηγικές και φιλόδοξη νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Όμως οι πολιτικές αυτές χρειάζονται ισχυρά μέσα και επίσης στήριξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτά, αυτό και ο οργανισμός του, τον οποίο συζητούμε, έχουν συμβάλει τα μάλα στην υλοποίηση της νομοθεσίας σε σχέση με ε, τι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα, κυρίως με τη στήριξη καινοτόμων ε, προγραμμάτων. Συγκεκριμένα δραστηριότητες όπως η περίπτωση των ε, νησιών και η περίπτωση των ε, φορέων τοπική αυτοδιοίκηση είναι σημαντική μοχλή στήριξη. Αυτό λοιπόν ε, προωθεί και την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή ώστε να εξασφαλίσει μια περίοπτη θέση για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκή ευθύ ενέργεια στην Ευρώπη στα πλαίσια του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου από το 2014 έω το 2020. Έπειτα, πώς σκοπεύει να βελτιώσει το επόμενο πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θεσμικώς πώς θα καλυφθεί το πρόγραμμα αυτό και στο πλαίσιο του ορίζοντα του 2020. Επίσης, τι κονδύλια θα το αποδοθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βότσον για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί καλύτερα όταν με λίγα χρήματα συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές και άλλους οργανισμούς για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. και όταν εκτελεί προγράμματα σε τομεί προτεραιότητας. Ε, το πρόγραμμα Εφής Ενέργεια και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία είναι εξαιρετικά παραδείγματα αυτού που μόλι προείπα για την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματο. Θα καταλαβαίνει λοιπόν η Κομισιόν τι ανησυχίε των βουλευτών όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχουν σχέδια διακοπή ενό προγράμματο που ενθαρρύνει του πολίτε να χρησιμοποιούν πιο συνετά την ενέργεια και βοηθούν την Ένωση να ανταποκριθεί στην εκπλήρωση των στόχων του Κιώτο. Η Κομισιόν λέει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τομέα αυτό. Αλλά ε, θα έπρεπε αντίθετα να ενισχυθεί αυτό το σκέλος στα επόμενα προγράμματα. Ο Επίτροπος Έτιγκερ χθε έλεγε ότι ίσως ε, πάει στον ορίζοντα 2020 το πρόγραμμα για την ευφυενέργεια. Θα υπάρχει όμως ένα ε, πρόγραμμα συγκεκριμένο, ιδιαίτερο. Θα έχει την προβολή που είχε αυτό το πρόγραμμα μέχρι τώρα. Θα κινητοποιηθεί η κοινότητα των πολιτών, θα υπάρξουν δεσμεύσει όπω αυτέ που είχαμε μέχρι τώρα. Όπω είπε και η κυρία Καρβάλιο, Υπάρχει το μέσο ε, για την ενεργειακή τοπική βοήθεια. Με πολύ μικρές επενδύσεις υπήρξαν σημαντικοί πόροι που βοήθησαν στην ενεργειακή απόδοση, για τη βελτίωση της ε, κοινωνικής στέγασης, για το σχεδιασμό ενεργειακά φιών κτηρίων μεταξύ άλλων, για την βελτίωση της ανανεώσιμης πηγής, ε, ανανεώσιμης ενέργειας και τη συμπερίληψή της στο δίκτυο Αποκεντρωμένε δραστηριότητε χρειάζονται λοιπόν για να προωθηθεί η εξοικονόμηση ενέργεια και ανανεώσιμε πηγές. Και το πρόγραμμα αυτό βοηθάει πολύ προ αυτή την κατεύθυνση. Ουσιαστικά αυτό που ρωτούμε είναι το εξή. Ε, σε ό,τι αφορά τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, η Κομισιόν πώ έχει χάσει το δρόμο τη, γιατί θέλετε να δώσετε χρήματα στα δίκτυα διανομή φυσικού αερίου προ όφελο εταιριών που ήδη βγάζουν δισεκατομμύρια κέρδο και γιατί δεν βάζετε αυτά τα χρήματα αντίθετα σε ένα όραμα που είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης ενεργειακά αποδοτικής, που μπορούμε να ε, μειώσουμε μέχρι το 2050 κατά 80% της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο λόγος στον κύριο Τούρμες για μισή λεπτά. Κύριε Λεβαντόφσκι, εγώ δεν ανησυχώ. Εξοργισμένος είμαι, όχι με εσάς προσωπικά, αλλά με εκείνους στη Γενική Διεύθυνση Έρευνα και Γενική Διεύθυνση Ενέργεια που αυτό το καιρό καταβάλουν μια προσπάθεια, ένα από τα πιο χρήσιμα προγράμματα που είχαμε ποτέ στο προπολογισμό να το καταργήσουν χωρίς αντικατάσταση. Μελέτες για αιωλικά πάρκα στη Βόρεια Θάλασσα. Κατάρτιση ε, υπαλλήλων στα κράτη-μέλη για την οδηγία για τα κτίρια. Αρχιτέκτονες και ε, μηχανικοί καταρτίζονται για το πώς ε, χτίζουμε τα καινούργια κτίρια. Δίκτυα μεταξύ προοδευτικών δημάρχων στην Ευρώπη και θα μπορούσα να συνεχίσω τον κατάλογο. Γιατί όλα αυτά τώρα θα πρέπει να καταστραφούν, για ποιο λόγο. Και αν η κυρία Γκέγενκριν και ο κύριος Ότιγκερ δεν έρθουν με συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχέδιο εμείς ως βουλευτές θα αναγκαστούμε να ξαναφέρουμε το παλιό ε, πρόγραμμα SIP καινοτομίας και ε, ανταγωνισμού και να το ξαναφέρουμε για το 2020 ε, ως ξεχωριστό ερευνητικό πρόγραμμα και καλά οργανωμένο πρόγραμμα καινοτομίας. Οι παρόντες συνάδελφοι γνωρίζουν πόσο μας ενδιαφέρει αυτό το πρόγραμμα και περιμένουμε και από την κυρία Γκέγγενκρουν και από τον κύριο Ότιγκε συγκεκριμένη απάντηση και γραπτή παρακαλώ και όσο γίνεται σύντομα. Αυτή η κατάργηση του προγράμματος για την ευφύ ενέργεια στην Ευρώπη είναι δηλητήριο αυτή τη στιγμή που προσπαθούμε και πρέπει να κερδίσουμε ε, τους Ευρωπαίους πολίτες. Εκείνοι που είναι ε, κινητοποιημένοι υπέρ τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερχόμαστε και τους ε, αποκρούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για δύο λεπτά η κυρία Ριέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η δική μου πολιτική ομάδα πάγια υποστήριζε και στεναρά την αύξηση του προπολογισμού για την έρευνα, για την ανάπτυξη αηφόρου ενεργειακής τεχνολογίας και θα συνεχίσει να το πράττει ε, στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Αλλά για να μπορέσουν τα αποτελέσματα της έρευνας να συμβάλλουν στην πολιτική μας για την ενέργεια, ε, ε, εξοικονόμηση ενέργειας και ανανεώσιμες, θα πρέπει να συνοδεύονται και από άλλα μέτρα, πάρα πολύ σημαντικά επίσης Μέτρα στήριξης σε δράσεις που στοχεύουν στο να διεισδύουν οι νέες τεχνολογίες στην αγορά και επίσης μέτρα για να αρθούν τα μη τεχνολογικά εμπόδια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγχυση ε, και να εμποδίσουν ε, τις τοπικές επενδύσεις στην κατάρτιση και τη ε, συμμετοχή των ε, τοπικών φορέων, όπως είναι το Σύμφωνο των Δημάρχων των ε, Ευρωπαϊκών Νήσων. Είναι ε, πολύ αξιόλογη η πρωτοβούλια που γίνεται. Έχουν γίνει πολλές αξιολογήσεις και το πρόγραμμα διακρίθηκε από την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν εδώ και τώρα να ξεκαθαρίσω ότι η δική μου πολιτική ομάδα υποστηρίζει τη συνέχιση του προγράμματος, τους στόχους του και ε, ε, τη ε, ισχυρή χρηματοδότηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πάξας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πρόγραμμα Εφής Ενέργεια για την Ευρώπη είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις, για τους ε, ενδιαφερομένους, ε, για τις πόλεις, να κάνουν διάφορες μελέτες για ε, πιθανές αλλαγές ε, και την νοτομία. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός για την καταπολέμηση ε, της κλιματικής αλλαγής και για την καλύτερη αξιοποίηση των ενεργειακών μας πόρων. Αν όμως θέλουμε να μιλάμε πραγματικά για ευφυή ενέργεια, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Αιωλική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, η υδροελεκτρική ενέργεια. Εναλλακτικέ πηγέ με δύο λόγια και εκεί να στοχεύουν όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Κανονικά εκεί θα πρέπει να υποστηρίζουμε τι επενδύσει και όχι στι ε, παλιέ ε, τεχνολογίε. Οι ανανεώσιμε είναι το μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε νέα προγράμματα, τολμηρά ας πούμε ενέργεια από υδρογόνο. Αυτές είναι οι μορφές ενέργειας. Πυρηνική ενέργεια, νέας γενεάς όμως. Από τις δικές μας αποφάσεις θα εξαρτηθεί το μέλλον του πλανήτη. Σε 200 χρόνια από τώρα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε σήμερα με αυτά τα θέματα και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις γι' αυτό. La parola al Ευχαριστούμε. Λόγω στον Επίτροπο, τον κύριο Λεβαντόφσκι. Thank you, Mrs. President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλα τα ερωτήματα, όλα τα σχόλια εξέφραζαν βαθιά ανησυχία για το μέλλον ενός προγράμματος που συνέβαλε πάρα πολύ συνεργική απόδοση και στην ανανεώσιμη ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Παραμένει δέσμευση, θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό, και θα ενισχυθεί και υπό οικονομικούς όρους στο μέλλον. Τα βασικά επιχειρήματα έχουν τεθεί επιτάπητος. Δηλαδή, χρήση, συμπολή προστιθέμενη αξία του προγράμματος εφής ενέργεια. Δεν θέλω να τα επαναλάβω αυτά τα επιχειρήματα, αλλά αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν είναι υποκειμενική εντύπωση μόνο. Τεκμηριώνεται, επιβεβαιώνεται και από εξωτερική αξιολόγηση, εξωτερική αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία είναι και πρόσφατα ε, και λέει, και θα το παραθέσω μεγάλη ικανοποίηση, ότι είναι και χρήσιμη και σημαντική γιατί ανταποκρίνεται σε προβλήματα και ανάγκες που σχετίζονται με τη βιώσιμη ενέργεια. Το πρόγραμμα ξέρετε ότι στήριξε περίπου 500 project, εκ των οποίων το 50% αφορούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι εδώ απαντώ στον κύριο Πάξας που εξέφρασε τη σχετική ανησυχία. Πραγματικά ένα υπόδειγμα ε, χρησιμότητας ε, προγράμματος ε, ευρωπαϊκού. Βέβαια, δεν μας ενδιαφέρει τόσο το παρελθόν και το παρόν όσο το μέλλον. Η απάντησή μου είναι εξής. Πολλούς στόχους πρέπει να πετύχουμε. Ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ένα. Πολύ σοβαρό θέμα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να απαντήσουμε και στο ζήτημα της αλληλεγγύης και της ενεργειακής ασφάλειας. Αυτό ήταν πάρα πολύ απτό το 2009, όταν και υπήρχε, έκλεισαν οι στρόφικες από τη Ρωσία προς την Ουκρανία. Και θα πρέπει να διασκεδάσουμε τις ανησυχίες θα πρέπει τους σπόρους μας να τους κατανείμουμε έτσι ώστε ναι με να αποσκοπούμε στην ε, ανάνωση μας πηγές ενέργεια, στην ενεργειακή απόδειξη αλλά και στα δίκτυα που συμβάλλουν και αυτά στην ενεργειακή ασφάλεια και στην αλληλεγγύη. Σε μια Ήπειρο που εξακολουθεί να εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τρίτες χώρες και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτά τα μονοπόλια. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας 100% αλλά πριν έρθω στην αίθουσα ε, μελέτησα αυτό το θέμα και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και συνέπεια μεταξύ ε, της ενημέρωσης των αγορών και της έρευνας και ανάπτυξης. Έτσι θα υπάρχει συγκεκριμένη συνιστόσα στο νέο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας του mainstreaming, της συμπερίληψης της, ε, διά, της ε, διάστασης αυτής σε όλες τις δράσεις μας. Στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, όπως τον αποκαλούμε. Ξεκίνησε ο αρμόδιος στον τον προπολογισμό. Δεν μιλάμε για μεγάλο ποσό, συμφωνώ. 743 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σαφής όμως η επίπτωση της μόκλευσης των χρημάτων αυτών. Άρα βλέπουμε εδώ πράγματι ένα παράδειγμα του πώς μπορούμε να πετύχουμε πολλά με λίγα χρήματα. Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει ε, να ενισχυθούν αλλά ξέρουμε ότι ο προπολογισμό δεν θα είναι αυξημένο. Το πώ θα γίνουν όλα αυτά θα το δούμε με μεγαλύτερε λεπτομέρειε το 2012. Αλλά θα ενισχυθεί αυτή η συνιστόση και είναι ένα από τα λίγα, από τα λίγα κονδύλια του προπολογισμού του 2012 που θα αυξηθούν. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε πάγωμα των κονδυλίων. Σε πραγματικές σταθερές θέλουμε να ε, έχουμε τον ε, προϋπολογισμό του 2012. Αυτή είναι η βασική αρχή. Έχουμε όμως το πρόγραμμα Horizon 2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 30 Νοεμβρίου. Θα τις γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες αργότερα, άρα δεν μπορούμε τώρα να έχουμε μια πιο αναλυτική συζήτηση. Όταν θα έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας μπορούμε να κάνουμε αυτή την πιο αναλυτική συζήτηση και σε ό,τι αφορά τον εκτελεστικό οργανισμό ανταγωνιστικότητα και καινοτομία. Και πάλι εδώ έχω να σα πω ότι η εξωτερική αξιολόγηση πολύ ξεκάθαρα έδειξε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο οργανισμό. Άρα ο ρόλο αυτού του οργανισμού και οι σχετικέ δραστηριότητε θα πρέπει να ενισχυθούν. Δεν είναι η δική μα εντύπωση. Έχουμε την εξωτερική αξιολόγηση. Και για το πρόγραμμα Εφής Ενέργεια, το δεύτερο αυτό πρόγραμμα, και για τον Οργανισμό Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας. Άρα και τα δύο θα πρέπει να τύχουν ε, καλύτερης ε, οικονομικής υποστήριξης μέσα στο ορίζοντα 2020. Εγώ αυτά έχω να πω, αλλά δεν είναι λόγια μόνο αυτά που λέμε. Είναι και στην πράξη αποδεδειγμένο ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Με αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ξεκινάει η συζήτηση με τους αγορητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων ξεκινώντας με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με την κυρία Ντελ Καστίγιο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, πιστεύω ότι η εξήγηση που δώσατε ήταν πολύ λογική και γεμάτη κοινή λογική. Παρόλες αυτές τις εξηγήσει όμως, καμιά φορά αυτά έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλα επιχειρήματα εξίσου λογικά. Στο Κοινοβούλιο τώρα τι θέλουμε εμείς να κάνουμε. Να επιστήσουμε την προσοχή γιατί ένα μέσο που στέφθηκε με επιτυχία να μην εξαφανιστεί στο βωμό θεωρητικών ε, λύσεων που μπορεί θεωρητικά να είναι πιο αποτελεσματικές αλλά εν πάση περιπτώσει έρχονται να ακυρώσουν την ανάπτυξη ενός μέσου που πραγματικά συνεισέφερε στην ύπαρξη πολλών προγραμμάτων με απτά ε, αποτελέσματα και με την εξοικονόμηση ενέργειας και πολύ σημαντικά δεν θα τα αναφέρω όλα δράσεις όπως ε, το Green Light, το Solar Keymark και άλλα, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι είναι επιτυχημένα προγράμματα και βασίστηκαν σε ένα θεμελιώδη πυλώνα. Και αυτούς τους καιρούς κρίσης που ζούμε στην Ευρώπη είναι ακόμα πιο πολύτιμα και ο άξονας αυτός της καινοτομίας. Οι κοινωνίες που δεν επενδύουν στην καινοτομία και στην κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής τους σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να επιβιώσουν σε μια τόσο ανταγωνιστική παγκόσμια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν το μέσο αποδείχθηκε και χρήσιμο για την ανάπτυξη της καινοτομίας στην ενέργεια. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε, ταπεινά επιμένουμε ένα τέτοιο μέσο να μην χαθεί να μην εξαφανιστεί. Θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να δούμε τι μοίρα θα έχει αυτή η υπόθεση, αυτό το μέσο για την FNA για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τη συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κ. Φανπρέντ, για ένα λεπτό. Κυρία Φανπρέντ. Πρόεδρε, Ελπίζω να τα πείτε κύριε Επίτροπε και στο συνάδελφό σας, γιατί με την απάντηση που μας δώσετε δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αν θέλετε η ενέργεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία μας να είναι δεδομένη, τι χρειάζεται σαφής επιλογή. Και το 2050 να έχουμε ποντάρει τα πάντα στις ανανεώσιμες πηγές και στην ενεργειακή απόδοση. Δεν υπάρχουν πιο σημαντικοί στόχοι από αυτούς τους δύο. Γι' αυτό χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και αυτό θα πρέπει να το επομιστεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά χρειάζονται και προγράμματα όπως είναι η ευφυής ενέργεια. Γιατί, για να φροντίσουμε σε τοπικό επίπεδο, πραγματικά με μικρότερα ποσά, να γίνουν πολύ μεγάλα βήματα και πρωτοβουλίες να αναλυφθούν. Ο Επίτροπος συνεχώς μας μιλάει για την ενεργειακή απόδοση και για τους καρπούς που αποδίδει αυτή σε τοπικό επίπεδο. Αυτό θα πρέπει να είναι ο πυρήνας του προγράμματος. Υπάρχουν τα χρήματα ε, θα πρέπει να αφιερωθούν σε αυτούς τους στόχους. Αυτό θέλουμε από σας να μας πείτε. Ευχαριστούμε. Δεν βλέπω τον ε, κύριο Κούρσκι. Νομίζω ότι δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Σόζα Βάγνερ για 1,5 λεπτό για τους μη εγγεγραμμένους. Παρακαλώ. Λουθ. Φως, περισσότερο φως λέει ζητούσε ο Γκέτε όταν έφευγε από τη ζωή. Σήμερα ο ποιητής που ήταν και πολύ καλός διαχειριστής σίγουρα θα ε, το έλεγε διαφορετικά. Ε, αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση φωτός. Γιατί μια Ευρώπη φτωχή σε ενεργειακούς πόρους χρειάζεται να ξέρει να κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην απαραίτητη κατανάλωση που οθεί την οικονομία και τη σπατάλη. Η σπατάλη ακριβώς θα πρέπει να χαλιναγωγηθεί. Γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε δραστική αλλαγή στην οτροπία και στις συνήθειες πολλών Ευρωπαίων πολιτών. Αναλύοντας την οικονομική κρίση ζητούμε και λιτότητα αλλά και κίνητρα για την ανάπτυξη. Λοιπόν, <clears throat> κανείς ή λίγοι τομείς προσφέρονται καλύτερα από τον ενεργειακό για να γίνουν αυτά τα ωραία λόγια πραγματικότητα. Μπορούμε να συνδυάσουμε και την τον περιορισμό της πατάλης και τις επενδύσεις. Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υποδομών που είχα την τιμή να παρουσιάσω την έκθεση ε, στο Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει πιο συγκεκριμένες προσπάθειες από ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα, διότι θα ενισχύσει αυτό τη σπονδυλική στήλη της Ευρώπης. Μόνο μία ισχυρή και καλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, ε, Πολιτική για την Ενέργεια συγγνώμη, ε, μπορεί να επιτρέψει στην Ευρώπη να προχωρήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ό,τι ε, κάνει προς την κατεύθυνση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ευπρόσδεκτο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Και τώρα οι λοιποί ο αγορτές. Ξεκινούμε με τον κύριο Μετσαρός για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην καινοτομία και να έχει μια ενεργειακή πολιτική και έναν εφοδιασμό αηφόρο. Η ρωσική κρίση του φυσικού αερίου, η πυρηνική καταστροφή ε, στη Φοκουσίμα και η εξάντληση των ορυκτών ε, πόρων ε, καθιστούν επίγουσα την ανάγκη να αστραφούμε αλλού. Το πρόγραμμα Εφής Ενέργεια για την Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει τα θεμέλια για μια καθαρή αηφόρο ενέργεια για τις επερχόμενες γενναίες και για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα προωθούνται πηγές και μείωση των ε, αέριο του θερμοκηπίου. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να προωθηθεί η έρευνα και η παιδεία. όλα αυτά λοιπόν το πρόγραμμα δυστυχώς ε, δεν είναι εξασφαλισμένο για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Γι' αυτό θα παρακαλούσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να εγγυηθεί αυτή την συνέχιση. Παρά τα συμβάντα στη Φουκουσίμα, Κατά την άποψή μου η πυρηνική ενέργεια ε, ανήκει στις ευφυείς πηγές ενέργειας διότι μπορεί να είναι και καθαρή ε, και ε, ασφαλής και ουδέτερη ως προς την εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα και στο ίτερ γίνονται πειράματα για αντιδραστήρες σύνδεξης που θα είναι αντιδραστήρες του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η επιτυχία του προγράμματος, το οποίο συζητούμε, μας δείχνει σαφώς ότι θα πρέπει να συνεχίσει. Υποστηρίζω λοιπόν την εξακολούθησή του και θα πρέπει να προβληθεί ακόμη περισσότερο στο πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο μάλλον ορίζοντας 2020. Αυτό που πρέπει να υποθεί ευθύ εξ αρχή είναι ότι θα πρέπει και εμεί το πρόγραμμα ευθύου ενέργεια να το διαδώσουμε περισσότερο στα νέα κράτη-μέλη. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση στο πρόγραμμα και αυτό πρέπει να γίνει προτεραιότητα, διότι πολλά κράτη-μέλη δεν συμμετέχουν ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν να τα παροτρύνουμε. Επίση, η καλύτερη πληροφόρηση για τα υπέρχοντα προγράμματα και του τρόπου που θα μπορούσε κανεί να έχει πρόσβαση στα κονδύλια για τη βελτίωση της συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν από την άποψη της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κόβαξ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρόγραμμα Εφής Ενέργεια είναι καταπληκτική πρωτοβουλία και αυτό το, δεν το λέω εγώ, το λένε αξιόπιστες πηγές. Πραγματικά είναι χρήσιμο για την Ευρώπη, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της, για την αηφορία. Ορισμένοι μάλιστα λέγουν ότι ε, μέχρι και οι φτωχοί Κινέζοι στραμμένα τα βλέμματά τους στην Ευρώπη ε, και ε, γεμάτη θαυμασμό μας παρακολουθούν. Προσέξτε όμως γιατί μπορεί να γελάνε μαζί μας, όχι να μας θαυμάζουν. Ε, γιατί βρισκόμαστε σε ένα πλοίο που βουλιάζει και θα πρέπει επιγόντως να το εγκαταλείψουμε. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο ασθενής. Με αυτή θα πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα και μετά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μόνο 2% του πληθυσμού μπορούν να πληρώσουν ε, την ακριβή ανανεώσιμη ενέργεια και το υπόλοιπο 98% τι γίνεται. Τα πυρηνικά εργοστάσια, εκεί επενδύει η Κίνα και η Ευρώπη όχι. Τελικά με το κερί θα φωτιζόμαστε στο μέλλον. Grazie. Σας ευχαριστούμε η κυρία Γιασλοβιέτσκα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ. Ένας από τους βασικούς στόχους στρατηγικής ε, για το 2020 είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι επίσης ε, η πρόθεση πράσινων τεχνολογιών δύσκολο θα είναι με την παρούσα κρίση να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, οπότε αυτό το μέσο ευφύης ενέργεια Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η λειτουργία του μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι αυξήθηκε η ενεργειακή απόδοση, προωθήθηκαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Υπήρξε μια ανταλλαγή, αν θέλετε, μεταξύ επιστημών και επιχειρήσεων και γι' αυτό και το νέο πρόγραμμα πρέπει να ε, επεκταθεί και να ανοίξει προς ε, νέα προγράμματα, νέες ε, πηγές, νέους πόρους. Και αυτό θα, επιτρέψει σε χώρες που απαιτούνται αλλαγέ να μπορέσουν να μειώσουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ο νέος ενεργειακός πόρος θα μας δώσει ανεξαρτησία είναι το σχιστολιθικό αέριο το οποίο έχει ανακαλυφθεί στην Πολωνία. Το θέμα είναι βέβαια οι στόχοι να μπορούν να ε, αξιολογούνται με τη συνεργασία βέβαια ειδικών ε, και των αρμόδιων εκτελεστικών οργανισμών. Έχουμε δει τέτοια θετικά παραδείγματα και καλό θα ήταν να μεταφερθούν και σε άλλους τομείς για να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα δράσεων και πιο βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Τσόγκ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί Πρόεδρε και ε, Επίτροποι, έχουμε τη στρατηγική 2020 για την Ευρώπη, έχουμε την ευφύη ενέργεια, έχουμε και εκτελεστικό ε, οργανισμό και διευκολύνσεις. Και τώρα μας λέτε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι όλα αυτά να καταργηθούν. για να φύγουμε από τους στόχους μας με τον πιο ακριβό τρόπο. Αυτό που μας χρειάζεται είναι να βελτιωθεί η ε, ενεργειακή απόδοση, η αποτελεσματικότητα στην Ευρώπη, να συμμετέχουν περισσότερες μικρομεσαίες. Αυτό θέλει το Κοινοβούλιο, συζητώντας ε, για όλα αυτά τα προγράμματα και τους επόμενους ε, μήνες. Ευχαριστώ κύριε Σπυρίλο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι, το πρόγραμμα e ευφυής ενέργεια είναι από τα κοινοτικά μέσα εκείνο που έχει τη μεγαλύτερη ε, επιτυχία ε, από όλα τα προγράμματα. Ε, εποφελούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μην μιλήσω για την προστιθέμενη αξία που έδωσε το ίδιο το πρόγραμμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Ανησυχώ κι εγώ, όπως και οι συνάδελφοί μου, για το μέλλον του προγράμματος, το οποίο διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στις δράσεις και στην ευαισθητοποίηση, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, κάνει ό,τι μπορεί για να συνεχιστεί το πρόγραμμα, γιατί η διακοπή του θα ε, είχε θα επέφερε απογοήτευση. Παρακαλώ, υπολογίστε και τη χρηματοδότηση και από πού θα βρεθεί. Ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγο στου αγορητέ με τη διαδικασία Κάτσδια, ξεκινώντα με τον κύριο Κέλλη. Παρακαλώ. Το περασμένο Σαββατοκυριακό διαπιστώσαμε πω είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε οτιδήποτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εξοικονόμηση ενέργεια και την αποδοτικότητα, προφανώ χρειάζεται πολλή χρόνο για να επιτύχει κανεί του στόχου του. Βεβαίω, η επιτυχία του προγράμματο ευθύς Ενέργεια για την Ευρώπη είναι κάτι που δύσκολα επαναλαμβάνεται από την πείρα μου. με με το πόσο αριθμ, τι μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, πόλεων, πολιτών έχουν έρθει σε μένα με προγράμματα, προγράμματα σχεδιασμένα ώστε να πραγματοποιηθούν εξοικονομήσεις ενέργειας και να βελτιωθεί η υποδοτικότητα βάσει νέων α, πλαισίων. Το νέο πρόγραμμα λοιπόν θα πρέπει είτε να εξακολουθήσει είτε να καλύπτεται από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με την ε, τοποθέτηση της Επιτροπής χτες, σε συνεδρίαση Επιτροπής, και όσα ακούσαμε σήμερα, βλέπουμε ότι χρειάζεται ένα συνολικό πακέτο που να διασφαλίζει ότι όλα αυτά μπορούν να συνεχιστούν. Ότι η, εξοικονό... η μείωση των εκπομπών κατά 80% με το 2015 είναι ένα στόχο που μπορεί να επιτευχθεί. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαγκίνε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι πήρε το μήνυμα η Κομισιόν ότι εμάς μας αρέσει το πρόγραμμα, είναι απλό, έχει αποτέλεσμα. Τουλάχιστον λοιπόν Θέλουμε ε, οι στόχοι να επικυρωθούν και σε, να συμπεριφθούν σε μελλοντικά προγράμματα. Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δεν φτάνουμε τους στόχους ε, της ενεργειακής απόδοσης και καθυστερεί αλλαγή της ε, κοινή γνώμη που θα έπρεπε να δεσμευθεί προ αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το, τον ορίζοντα 2020, αυτή η έννοια περί φιού ενέργειας είναι κάτι που ίσως ε, χαθεί μέσα στο ευρύτερο αυτό πρόγραμμα. Εξού και θα πρέπει να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ολοκληρώνοντας να πω ότι γιατί προσπαθούμε να κολλήσουμε κάτι που δεν έχει σπάσει. Θα ήθελα να δώσετε αυτό το μήνυμα στους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάτουλα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Το πρόγραμμα Εφής Ενέργεια Ευρώπη πραγματικά αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την εφή χρήση της ενέργειας στον τομέα των μεταφορών, ενεργειακή απόδοση κτηρίων, βιομηχανική κατανάλωση και ούτω καθεξής. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο αν θέλουμε να μειώσουμε τις εκπομπές ρήπων, να εκπληρώσουμε τους φιλοδόξους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιες πρωτοβουλίες θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ επιτυχής, ιδίω αν ξεκινούν από το τοπικό επίπεδο. Πρέπει να υπάρχει όμως και καλύτερη ενημέρωση και καλύτερη και περισσότερη συμμετοχή των αρχών ενεργειακές λύσεις για ενεργειακά βιώσιμα κτίρια, πιο καθαρά αυτοκίνητα, προγράμματα αστικής κινητικότητας. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία προωθούν την αηφορία και την ενεργειακή απόδοση στα αστικά κέντρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Τράπεζα Επενδύσεων, την Κομισιόν, νομίζω ότι αν βοηθήσουν και οικονομικά θα βελτιώσουν τα προγράμματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μέρκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, εκτιμώ τις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλούστευση, για σαφείς στόχους, αυτό που λέτε mainstreaming, αλλά δεν χρειάζεται να επανεφεύρετε τον τροχό. Όταν λειτουργεί κάτι καλά, λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να το αλλάξουμε και να το επαναφέρουμε με άλλο τρόπο, με άλλο όνομα. Αφήστε το στην ησυχία του. Το πρόγραμμα Φύση Ενέργεια για την Ευρώπη λειτουργεί, αποδίδει, το είπατε, φτάνει στους πολίτες, φτάνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χρειαστήκαμε τόσο καιρό για να φτάσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο κοντά στους πολίτες. Το είπε χθε ο συνάδελφός σας, Ότιγκερ, ότι το πρόγραμμα ε, έχει σχεδιαστεί και θα μας ενημερώσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αργότερα. Ε, γιατί λοιπόν άσκοπα να κάνετε αυτές ε, τις ενέργειες. Και μπορείτε να μας πείτε πού θα ενταχθεί ακριβώς αυτό το πρόγραμμα, ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός του, ποιοι θα είναι οι στόχοι του, τα μέσα, πώς θα διευρυνθεί και τι θα γίνει στο μέλλον και στο επόμενο πολιετές ε, πρόγραμμα και στο πρόγραμμα ορίζων θα το έχουμε. Κατά τα άλλα θα ήθελα να πω ότι και το Horizon 2020 είναι καλή προσπάθεια για την έρευνα, αλλά ακριβώ αυτά τα προγράμματα που είναι τόσο πρακτικά και συμμετέχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ λίγα, είναι πολύ πολύτιμα και θέλουν την προσοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου, νομίζω δεν βρίσκεται στην αίθουσα. Οπότε να δώσω το λόγο στον κύριο Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το πρόγραμμα Ευφύης Ενέργεια για την Ευρώπη ε, δημιουργήθηκε το 2003 και γέννησε έντονο ενδιαφέρον. Μέχρι σήμερα ε, χρηματοδοτήθηκαν και υλοποιήθηκαν από 200 σχέδια και έργα για για την κοινωνία της γνώσης, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμμερίζομαι και εγώ τις αγωνίες για το μέλλον του προγράμματος αυτού. Θα πρέπει στα πλαίσια της επόμενης προγραμματικής περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών να διατηρηθεί για να μπορέσουν να συμμετέχουν τα ερευνητικά αισθητούτα και να ε, ε, δημιουργηθεί καινοτομία στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άλβες. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επενδύσει στην ε, οικονομία της γνώσης και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να αναζητήσουμε την ανεξαρτησία μας από το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα κίνητρα και τις επενδύσεις μας. Εδώ έχουμε ήδη κάποιες δοκιμές για παραγωγή δεοθερμική ενέργειας από ηφαιστειακέ πηγές τις Ασόρε. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε στι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διότι πολλές φορές η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 50% διασφαλίζεται από γεωθερμικές πηγές. Αυτό σε ορισμένε περιοχέ και σε ορισμένε περιόδου του έτους, όπου εκεί θα μπορούσε να στραφεί κανεί στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Έτσι λοιπόν οι Ασόρε θα γίνουν το πρώτο νησί παγκοσμίω που θα είναι 100% τροφοδοτούμενοι από ανανεώσιμε πηγέ. Να ένα πολύ καλό παράδειγμα για το μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και την ευθύ ενέργεια. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Πάσκα. Ευχαριστώ πολύ για να καταφέρουμε να έχουμε μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να υπάρχει επαρκής ενέργεια. Αυτή τη στιγμή εξαρτώμαθε από εισαγωγές από την Ασία και την Αφρική. Δηλαδή δεν έχουμε στη διάθεσή μας ε, επαρκείς πηγές φυσικού αερίου και γι' αυτό θα πρέπει να ψάξουμε εναλλακτικέ πηγές. Και αυτό το πρόγραμμα ευφυής ενέργεια πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια πρέπει να βρούμε μοντέρνες, σύγχρονες λύσεις και να αναζητήσουμε νέες πηγές ενέργειας. Εκπνέει το πρόγραμμα, γι' αυτό πρέπει ευθύ αμέσω να διερωτηθούμε τι θα γίνει στο μέλλον αυτή την πρωτοβουλία μετά το 2013. Τι θα κάνουμε, πώς θα προχωρήσουμε και εγώ και οι συνάδελφοί. Κύριε Επίτροπε, πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να απαντηθεί αυτό το ερώτημα από την Κομισιόν. Ευχαριστούμε κύριο Σικέρσκι. Το πρόγραμμα που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενίσχυση για να βελτιωθεί και η ενεργειακή αποδοτικότητα για τους ενεργειακούς μας πόρους και για την προστασία τους θα πρέπει τα προγράμματα που θα εγκριθούν να καλύπτουν ένα μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας λοιπόν και της εξοικονόμησης ενέργειας θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη όθηση ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ χρειάζονται αλλαγές στο πρόγραμμα οι οποίες περιβαλλοντικώς θα πρέπει να είναι πολύ σωστά σχεδιασμένες ώστε και οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα να περιοριστούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μέρος της δέσμευσής μας για το μέλλον. Θα πρέπει οι λύσεις μας για την εξοικονόμηση ενέργεια να είναι εξυγχρονισμένες και βεβαίως να τρέξουμε και στις ανανεώσιμες πηγές. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τελευταία παρέμβαση από την κυρία Τσικάου. Grazie mille. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαστε υπέρ τη συνέχιση του προγράμματο Εφή Ενέργεια και στι μελλοντικέ μεσονομικέ προοπτικέ, γιατί το πρόγραμμα αυτό ενθαρρύνει τη δημιουργία εφιών ενεργειακών λύσεων. Για την περίοδο 2007-2013 έλαβε 713 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα παρέσχει 75% χρηματοδότηση στα επιλέξιμα προγράμματα. Έχουν χρηματοδοτηθεί λοιπόν πάνω από 500 project διάρκεια 2 έω 3 ετών και 8 με 9 συμμετέχουσε χώρε. Δηλαδή πάνω από 3.000 ήταν οι δικαιούχοι σε 21 χώρε. Για να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση βέβαια θέλουμε να πούμε ότι 250 project σε στους τομείς μεταφορών των ενεργειακών κτηρίων και τα λοιπά έχουν ξεκινήσει και για όλα αυτά θεωρούμε ιδιαίτερα ευεργετικές επιπτώσεις του προγράμματος εφής ενέργεια που χρηματοδότησε όλα αυτά τα προγράμματα. 476 προγράμματα φέτος με 328 σχολές από την Ευρώπη και από Κροατία, Νορβηγία έχουν ε, δρομολογηθεί και θα θέλαμε να Επιμείνουμε λοιπόν στη συνέχιση του προγράμματος αυτού και στο προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα Επίτροπος Λεβαντόφσκι. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, μου είπατε ότι θα πρέπει να πείσω για τη χρησιμότητα ενός προγράμματος, μάλλον καταφέρατε να με πείσετε για τη χρησιμότητα ενός προγράμματος, που είναι τόσο επιτυχημένο, που είναι αποδοτικός προς το κόστος, που έχει 713 εκατομμύρια ευρώ πρικοδότηση και τεράστιες επιπτώσεις ως προς τις βελτιώσεις των επιδοσεών μας στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, μιλήσαμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ακριβώς ανήκουν στους 3.000 ε, εταίρους μας, τους συνεργάτες του τους 3.500 συνεργάτες που θα μπορούσαν να βρεθούν στην κατηγορία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εδώ λοιπόν αυτό που έχω να δηλώσω προ το Ευρωκοινοβούλιο είναι ότι χάρη σε εσά αυξήθηκε ο προπολογισμό για το 2011 κατά 10 εκατομμύρια ευρώ και για το επόμενο έτο κατά 7,5 αυτό λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ε, πραγματικά δέσμευση ω προ το πρόγραμμα αυτό και αυτό εκφράζεται με συγκεκριμένε δημοσιονομικέ γραμμέ. Δεν θα εξαλειφθεί το πρόγραμμα αυτό. Μια δέσμευση δεν εξατμίζεται έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Ε, περιλαμβάνεται στους στόχους της στρατηγικής του 2020 και η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι μεταξύ των 7 τομέων προτεραιότητας της στρατηγικής μας για το μέλλον της Ευρώπης. Ωστόσο, θα πρέπει να ανταποκριθούμε και στην ανάγκη για ευθυγράμμιση των προγραμμάτων. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από όλες τις επισκοπήσεις, τις αποτιμήσει, τις αξιολογήσεις των προγραμμάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα χρειαστεί στο μέλλον λόγω των περιορισμών. Θα πρέπει να δαπανούμε όχι περισσότερα κονδύλια λόγω του κόστους που υπάρχει αλλά, και των δυσκολιών, αλλά πώ θα δαπανούμε καλύτερα. Δεν θέλουμε λοιπόν να εξαφανιστεί ένα πρόγραμμα που θα πάει τόσο καλά. Τώρα ποιο είναι το μέλλον του προγράμματος αυτού. Θα πρέπει να βρεθεί σε ένα συνεκτικό πλαίσιο που να διασυνδέει την έρευνα της επενδύσεις και την επικαιροποίηση της αγοράς με ε, ένα αυξημένο χαρτοφυλάκιο με τον ορίζοντα του 2020 θα πρέπει να περάσει από τα 50 στα 80 εκατομμύρια ευρώ ενώ η συνιστόσα της ενέργειας θεωρείται ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια αυτή που παράγεται μέσω του προγράμματος αυτού. Δεν μπορούμε λοιπόν να αμελήσουμε την διάσταση της ασφάλειας, αυτή την ε, ήπειρο, της ενεργειακής δηλαδή ασφάλειας, που τα ερχόμενα χρόνια θα εξαρτηθεί και από το τι θα στο πρόγραμμα του Ορίζοντα το 2020. Θα πρέπει λοιπόν να επιζητούμε καθαρή και αποδοτική ενέργεια, δηλαδή ευφυή ενέργεια. Αυτό σημαίνει ευφυή ενέργεια. Δεν ε, μπορούμε να ξεχνάμε αυτό το ειδικό στοιχείο ε, της ενεργειακής συνιστώσας. Θα πρέπει αυτή η δέσμευσή μας και σε χρηματικού ε, όρου, δηλαδή από την άποψη των κονδυλίων, να είναι σαφή. Θα πρέπει να ξέρουμε βέβαια πόρου για την ευφυή ενέργεια και για τι ανανεώσιμε πηγέ και για την ενεργειακή υποδοτικότητα. Όπω θα γνωρίζετε κατά πάσα πιθανότητα, αυτό μεταξύ των προτεραιοτήτων των διαφορετικών ταμείων βρίσκεται πολύ ψηλά. Μεγαλύτερο κονδύλι και Έχουμε και τις ε, περιοχές της ενδιάμεσης κατηγορίας, κάτω του 90% του ε, μέσου όρου ΑΕΠ, κατά κεφαλή ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε δηλαδή για ένα συνδυασμό στόχων. Η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι το νούμερο ένα στα διευθυντικά ταμεία και σε αυτόν τον τομέα και ακριβώς σε αυτήν την κατηγορία περιφερειών στην Ευρώπη. Εδώ λοιπόν δεν θα μιλήσουμε αυτό το στόχο. Τώρα θέλουμε μία θέση για την ευθύ ενέργεια και στο πολιετές δημοσιονομικό πλώσιο. Θα θέλαμε ίσως περισσότερο και από ένα δί. Δεν μπορώ να πω εάν θα υπάρξει τέτοιο ποσό, όμως το χαρτοφυλάκιο διαρκώς διωγγώνεται. Υπάρχει λοιπόν και οικονομική δέσμευση και προβολή του στόχου και αυτό θα φανεί και στον ορίζοντα του 2014-2020. Ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ σαφής, προκειμένου να καθορίσουμε το μέλλον, να καθορίσουμε τους όρους του παιχνιδιού σε αυτό το σκέλος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε και τώρα στην ημερήσια διάταξη η έκθεση ΣΒΑΜ για την πολιτική ανταγωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δώσω αμέσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σφαμπ, για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Διπρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, καταρχά θα ήθελα